Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη Συμφωνία Προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, Υπουργό, τον κύριο Λοπές Καρίγκο. Έχετε το λόγο εξ του Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει το πρώτο ανθρώπινο δικαίωμα που είναι το δικαίωμα στη ζωή. Στην Αθήνα ήταν αυτό αποτέλεσμα, οι τρεις νεκροί ήταν το αποτέλεσμα βιαίων ενεργειών τις οποίες καταδικάζουμε κατηγορηματικά. Η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου, ξέρω του Συμβουλίου, θέλει να εκφράσει τα συλληπιτήριά του και την αλληλεγγύη της προς των θυμάτων και γι' αυτό προσυπογράφει τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. <clears throat> Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα από αυτά, όπως είπαμε, το δικαίωμα στη ζωή και στην σωματική ακυρεότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και, τα, και τις πολιτικές ελευθερίες. Όλα τα κείμενά της έχουν πάντα μια μόνιμη παραπομπή <clears throat> στις θεμελιώδεις αυτές ελευθερίες που περιλαμβάνει και αυτή η σύμβαση. Και η κορύφωση αυτής της διαδικασίας είναι η Συνθήκη της Λισαβόνης. Η Συνθήκη της Λισαβόνης, από τη μία πλευρά ενσωματώνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της Ευρώπης που έχει ένα χαρακτήρα δεσμευτικό νομικά και παράλληλα λέει για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει τμήμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κορύφωση αυτής της πορείας, αυτής της πολιτικής, νομικής και πολιτιστικής τροχιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που θέτει την χάρτα αυτή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο της νομικής προσωπικότητας και της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη, ώστε εν καιρό να μπορέσει να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αποδέχεται την δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Και έτσι αυξάνουμε τις εγγυήσεις προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και μια προσέγγιση, μια σύγκληση μεταξύ των νομικών πλαισίων των κρατών μελών σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ένομε τάξει που υπάρχουν σε κάθε μία από τι δημοκρατικέ χώρε τη Ευρώπη, οι οποίε σέβονται και προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη μία πλευρά και <clears throat> του νομικού της ένομης τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του πλαισίου τη Συμβουλίου τη Ευρώπη, που είναι ένα ευρύτερο γιατί το απαρτίζουν όχι μόνο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλε χώρε τη Ευρώπη που δεν είναι τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία σύγκλησης αυτών των ενόμων τάξεων και η κορυφωσή του θα είναι ακριβώ η υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει 17 Μαρτίου μια σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση αυτή. Το Συμβούλιο έχει πράξει έκτοτε ότι είναι δυνατόν για να μπορέσει να επιταχύνει την πορεία των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει μια ομάδα εργασία στο Συμβούλιο και που προσπαθεί να προωθήσει αυτέ τι διαπραγματεύσεις σε στενή σύνδεση με την Κομισιό. Το Συμβούλιο έχει λάβει σοβαρά υπόψη όλες τις εντολές αυτές που αναφέρονται στο πρωτόκολλο 8 που είναι το σημείο αναφορά σε νομικό επίπεδο, παραδείγματο χάρη την ενδεχόμενη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελεγκτικά όργανα τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η ανάγκη να προσαρμοστούν και να τύχουν σεβασμού οι αρμοδιότητε αυτών των οργάνων. Επίση, η δυνατότητα να υπάρχει ένα δικαστή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συμμετέχει επίση το κοινοβούλιο μα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη και επίση στην Επιτροπή των Υπουργών όταν ασκούνται ε, εγχειρήματα και καθήκοντα που έχουν να κάνουν με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, το Συμβούλιο έχει παρακολουθήσει προσεκτικά την ακρόαση, τι ακροάσει μάλλον που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο για τα θέματα αυτά και έλαβε πάρα πολύ προσεκτικά υπόψη τα επιχείρηματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κυρία ε, Γκάλ και τον κύριο Χαουραγή Ατόντο που ήταν εισηγητέ. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η εντολή διαπραγματεύσεων για θέματα τα οποία είναι πολύπλοκα και τεχνικά αυτή η εντολή προς την Κομισιόν για τη διαπραγμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010. κυρία Ρέντινγκ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνάδελφος Όλη Ρέν ήδη εξέφρασε την θέση και τα συλληπιτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ελληνική καταστροφή. Ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τη δουλειά μας, διότι αυτό θα είναι υψίστης σημασίας για την ολοκλήρωση του συστήματος προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ενώσεως και η προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ενώσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι κάτι που αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι επιλογή, είναι προορισμός. Όπως τόσο καλά το εξέφρασε μόλις τώρα και η Προεδρία. Αυτή η προσχώρηση είναι ένα μόνο από τα τέσσερα στοιχεία πολύ φιλόδοξων ε, πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα και πολύ ε, πλήρων πολιτικών ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη, μόνο τέθει σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων γίνεται δεσμευτικός, δεσμευτική νομικά. Και αυτή η χάρτα είναι η πιο σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κόσμο όσον αφορά πολιτική δέσμευση για την υλοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων νομική ασφάλεια και περιέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη σύμβαση. Το νόημα και το πεδίο εφαρμογή των δικαιωμάτων είναι τα ίδια όπως αυτά τη συμβάσεως, αλλά η χάρτα προχωρεί πιο πέρα, διότι, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται η τρίτη γενιά θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ακαλείται, δηλαδή προστασία δεδομένων, εχέγγια για, τα, για δεδολογικό κώδικα, για βιολογικά θέματα, κώδικα θεντολογικός και σωστή διοίκηση. Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τη χάρτα θα πρέπει πάντα να είναι τουλάχιστον εξίσου υψηλό όπως αυτό της συμβάσεως. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο υψηλό και προωθούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό θεωρείται ως προτεραιότητα του προγράμματος της Στοκχόλμης που καθορίζει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Και τρίτον, προβλέπεται η δημιουργία του νέου χαρτοφυλακίου δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια που δείχνει πόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδίδει σημασία στην ενίσχυση της δράσης αυτής σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέταρτον, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Σύμβαση θα εγγυάται ότι οποιοδήποτε άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα παραβιάσεως της συμβάσεως από θεσμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δύναται να προσφύγει κατά της Ενώσεως προσφεύγοντας στο δικαστήριο του Στρασβούργου υπό τους ίδιους όρους όπως εκείνοι που κάνουν καταγγελίες κατά των κρατών μελών σε, από πολιτική σκοπιά, αυτή η προσχώρηση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου το βασικό ρόλο που διαδραματίζει το σύστημα της συμβάσεως για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη σε μια διευρυμένη Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχωρώντας λοιπόν σε αυτή τη σύμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το σύστημα του Στρασβούργου. Βάζει το βάρος της πίσω από το σύστημα του Στρασβούργου. Είναι ένα σύστημα εξωτερικού δικαστικού ελέγχου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι τώρα θέτουμε τη νομική μας τάξη πλήρως και επισήμως σε αυτό τον έλεγχο. Αυτό βεβαίως θα αυξήσει την αξιοπιστία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και θα φανεί ότι είναι δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει και να προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα. Τα μέσα Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο εντολή διαπραγματευτική. Το πρωτόκολλο 8 της Συνθήκης της Αβώνας απαιτεί κάποιες ουσιαστικές εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχονται σε μια συμφωνία που σχετίζεται με αυτή την προσχώρηση, διότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νόμου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο λαμβάνει πλήρως υπόψη αυτές τις απαιτήσει. Ήθελα κυρία Πρόεδρε απλώς να αναφέρω δύο από αυτά τα στοιχεία. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εξουσίες της και αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως καθορίζονται στις συνθήκες δεν μπορούν να επηρεαστούν από αυτή την προσχώρηση. Και η συμφωνία προσχώρηση θα πρέπει αυτό να το αναφέρει ρητά, να το κάνει ξεκάθαρο. Παρομοίω, η προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε την κατάσταση που αφορά τα διάφορα μεμονωμένα κράτη-μέλη έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε τα πρωτόκολλα, τα σχετικά, ούτε τι επιφυλάξει. Οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπώ ότι η Συμφωνία προσχώρηση δημιουργεί υποχρεώσει σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις των συμβάσεων μόνο σχετικά με πράξεις και μέτρα που υιοθετούνται από τα θεσμικά όργανα ή φορείς της Ενώσεως. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει μια ομαλή ένταξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο σύστημα της συμβάσεως. Η ένταξη θα πρέπει να διατηρήσει τα ουσιαστικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Όμως, η ένταξη αυτή, η προσχώρηση θα πρέπει να πληρεί δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, όπως προανέφερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νόμου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί, διαφυλάσσοντας το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα προνόμια του μετά την ένταξη είναι σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν ενδιαφέρουσε ε, προτάσει ε, επί τραπέζης που έχουν σαν στόχο τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε περιπτώσει όπου η συμβατότη νομική πράξεω τη ενώσεω διακυβεύεται ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, άνευ ε, προδικαστικής διαδικασίας. Αυτές οι προτάσεις πιθανότατα μπορούν να σχεδιαστούν τι ούτω τρόπος, ούτως ώστε να μην απαιτούν τροποποίηση της συνθήκης και Πρόεδρε, θα πρέπει και αξίζει να γίνει προσεκτική ανάλυση και συζήτηση για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο και στα διάφορες, στις διάφορες ομάδες εργασίες του Συμβουλίου και γνωρίζω ότι η Ισπανική Προεδρία κάνει τα πάντα ούτω ώστε να προωθηθεί και να προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Δεύτερον, είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με την ιδιαίτερη κατάσταση της ενώσεως που είναι ξεχωριστό νομική προσωπικότητα με αυτόνομες εξουσίες που θα είναι αντισυμβαλόμενο μέλος μαζί με τα κράτη-μέλη και θα προσχωρήσει ένα μηχανισμό που αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό αλλά είχε σχεδιαστεί για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό περιορισμένος αριθμός τεχνικών και διαδικαστικών προσαρμογών ε, είναι κάτι που απαιτείται στη Σύμβαση όσον αφορά την ιδιαίτερη φύση του νόμου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως και του, του μηχανισμού που αφορά την επαφή των αντισυμβαλωμένων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αποκεντρωμένη εφαρμογή του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη. Μέσω αυτού του μηχανισμού το, η Ένωση θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις διαδικασίες σαν συμβαλόμενο μέλος ε, σαν διάδικος άμα δικάζεται ένα κράτο μέλο. Από θεσμική απόψεως ε, θα ήθελα να τονίσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ότι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να συμμετέχουν στους φορείς της συμβάσεως σε ισότιμη βάση με τους ε, εκπροσώπους άλλων συμβαλωμένων μερών. Τι σημαίνει αυτό ότι ένας δικαστής που εκλέγεται από κάθε συμβαλόμενο ε, μέρος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, δηλαδή κάθε νομικό σύστημα αντιπροσωπεύεται εντός του δικαστηρίου. Επίσης αντικατοπτρίζεται, το συλλογικό σύστημα εγγυήσεων που δημιουργείται από τη Σύμβαση, όπου κάθε συμβαλόμενο μέρος απαιτείται να συμμετέχει. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ε, ένα μόνιμο πλήρη δικαστή που θα εκλέγεται για την Ένωση και θα έχει το ίδιο καθεστώς και τις εξουσίες με τους ομολόγους του και θα παρεμβαίνει ενδεχομένως σε όλες τις υποθέσεις. Κυρία Πρόεδρε, ένας ad hoc δικαστής που παρεμβαίνει μόνο σε, περι... υποθέσεις που στρέφονται κατά της ενώσεως, που εμπλέκουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θα ήταν κάτι που θα αρκούσε. Όσον αφορά τη μέθοδο εκλογής του εν λόγω δικαστού, η κανονική διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση θα πρέπει να εφαρμόζεται και εδώ. Αυτό σημαίνει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη εκλέγει αυτό το δικαστή από κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ενδεδειγμένο αριθμό μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχει σε συνεδριάσει τη κοινοβουλευτική Συνελεύσεω όταν αυτή θα εκλέγει τους δικαστές για το δικαστήριο του Στρασβούργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές των Επιτροπών ΑΦΚΟ και ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Γιαρέγγι και την κυρία Σκολ, για την έξοχη συνεργασία όσον αφορά το θέμα αυτό και για την ακρόαση που διοργανώθηκε την Επιτροπή ΑΦΚΟ στις 18 Μαρτίου που πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Επίσης χαίρομαι που η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου έδωσε με ύψιστη προτεραιότητα στο χαρτοφυλάκι αυτό και έχω κάθε πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη μετά το καλοκαίρι και θα εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν διαπραγματευτή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα ενημερώνει πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τη σχετική διαδικασία. Κυρία Πρόεδρε, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται μια τέτοια μέρα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Ευρώπη και πόσο σημαντικά είναι για όλες όλε τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και είμαι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στι προδιαγραφέ που επιτάσσει η Σύμβαση. Αλλά η προσχώρηση, η ένταξη στη Σύμβαση σίγουρα είναι κάτι που θα αυξήσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και εννοώ τα δικαιώματα του κάθε ενός ανθρωπίνου όντω που ζει στην Ευρώπη. Κύριε Αντιπρόεδρε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων τώρα θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Από το, για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά έχει το λόγο. Πολύ κυρία Πρόεδρε, προσυπογράφω απόλύτω τι δηλώσει του Υπουργού κυρίου Λαούπε Γκαρίδο εκ μέρου τη Ισπανική Προεδρία, καθώ και τη Αντιπροέδρου κυρίας Ρέντινγκ και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ραμόν Χαουρεγκή και την κυρία Γκάλ για τι εισηγήσει του και τη δουλειά που πραγματοποίησαν η προσχώρηση της ευρωπαϊκής ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση ε, του συμβουλίου της ευρώπης και στα πρωτόκολλά της αποτελεί εφαρμογή της συνθήκης της λισαβόνας και διευρύνει την προστασία στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πολίτες της. διαμορφώνεται έτσι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτεται από την ομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του στρασβούργου ενώ ταυτόχρονα εκτός από την εξωτερική προστασία ε, η ευρωπαϊκή ένωση αποκτά έναν εξωτερικό φορέα προστασίας με διεθνή χαρακτήρα ενισχύοντας την αξιοπιστία της και έναντι τρίτων χωρών από τις οποίες συχνά αξιώνει στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων να σέβονται την ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. κυρία πρόεδρε η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες συμπίπτει σήμερα με τη δολοφονία τριών πολιτών εργαζομένων από ακραία και περιθωριακά στοιχεία στη χώρα μου στην αθήνα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον των μέτρων της κυβέρνησης που αφορούν στην οικονομική κρίση. θέλω εκτός από τη συντριβή και την οδύνη μου και εκ μέρους των συναδέλφων μου της μείζωνος αντιπολίτευσης στην ελλάδα να σημειώσω ότι η πολιτική μας παράταξη είναι αποφασισμένη να συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημοκρατίας και την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών. Κυρίες και κύριοι, σεβόμαστε τα χρήματα που μας δίνονται αυτή την κρίσιμη στιγμή από τους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Ως υπεύθυνο κόμμα θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την προστασία της ομαλότητας και την ενότητα του ελληνικού λαού απομονώνοντας τα ακραία στοιχεία που υπονομεύουν τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαννάκου. Τώρα εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, ο κύριος Γιαουρέγγι για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αν έπρεπε να συμπυκνώσω μονάχα σε μια ιδέα αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα, θα ήθελα να πω με μεγάλη σαφήνεια σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για πρώτη φορά θα έχουν ένα δικαστήριο το οποίο να εξασφαλίζει τα βασικά τους δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι των κρατών μελών όταν εξελίσσουν το κοινοτικό, όταν μεταγράφουν και εξελίσσουν το κοινοτικό δίκαιο. Η ιδέα είναι ότι το νέο αυτό δικαστήριο του Στρασβούργου θα εμφανιστεί ενώπιον των πολιτών ω εγγυητή του ότι το κοινοτικό δίκαιο και η εφαρμογή του ίδιου αυτού κοινοτικού δικαίου σε κάθε κράτο μέλο θα τηρήσει τι ελάχιστε εγγυήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι οι, οι ιδέε που βρίσκονται στον πυρήνα τη ευρωπαϊκή ιδέα που είναι ο ομφάλιος λόρος της ευρωπαϊκής κατασκευής, που είναι μια κατασκευή πολιτισμική που βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξιοπρέπειας των ατόμων και η οποία συμπυκνώνεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν μας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συγκεκριμενοποιήσει, όπως είπε και η κυρία Ρέντιν τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι η πιο εξελιγμένη τέτοια χάρτα που υπάρχει στον κόσμο και μας υποχρεώνει να την ενσωματώσουμε και να αποδεχτούμε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Αυτό θα εγκρίνουμε τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα. Θέλω να υπογραμμίσω όμως τη σημασία του γεγονότος ότι η Κομισιόν έχει προβεί σε ένα ταχύ και αποτελεσματικό έργο με την επίτευξη μιας, πρώτα, εντολής που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Ρέντιν για την αποτελεσματικότητά τη και επίση θέλω να ευχαριστήσω και την Ισπανική Προεδρία. Στην επόμενη Ολομέλεια του Μαου, <clears throat> εμεί θα εγκρίνουμε την έκθεση του, Κοινο... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και θέλω να σα ζητήσω να υπάρξει πληροφόρηση και παρουσία του Κοινοβουλίου σε μια διαπραγμάτευση που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Τώρα για δύο λεπτά επίση η κυρία Βίστρομ εκ τη Συμμαχία των Φιλελευθέρων. E η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στο ε, Δικαστήριο Δικαιωμάτων εδώ και πολύ χρόνο ήταν σχέδιο. Τώρα έχουμε συγκεκριμένη βάση για να γίνει αυτό. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση συνεπάγεται την ενίσχυση της προάστησης των δικαιωμάτων. Οι πολίτες της χώρας μας θα έχουν καλύτερη προστασία σε σχέση ε, και θα υπάρχει καλύτερο συντονισμός ε, στην ε, νομική πρακτική και στα δύο δικαστήρια. Με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόσπιση των δικαιωμάτων θα εγγυηθούμε την ανεξάρτητη τον ανεξάρτητο σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Είναι πολύ εύκολο, κυρία Πρόεδρε, να θεωρήσουμε ότι στην Ευρώπη είμαστε ελεύθεροι από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, πραγματοποιούνται σε άλλα μέρη του κόσμου. τα ε, μέλη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ε, νομοθεσία που διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία λόγου είναι ευρωπαϊκά δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται πάντα διότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου παραβιάζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αφήνουμε να γίνεται αυτό. Με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση με στόχο την ενίσχυση ε, και τη συμπλήρωση των ε, δικαιωμάτων των πολιτών είναι σημαντικό ε, το Κοινοβούλιο να νομοθετεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή διότι είναι γεγονό ότι στα κράτη-μέλη μας υπάρχουν, απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν για να ενισχύσουμε με πράξεις τα ωραία λόγια, τα ε, οποία λέμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να παρακαλέσω τους ε, συναδέλφους και τις συναδέλφους να σέβονται τον χρόνο, να τηρούν τον χρόνο που τους έχει ε, διανεμηθεί, γιατί έχουμε βαρύ πρόγραμμα μέχρι το βράδυ. Η κυρία Χαουτάλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι θεωρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν κάτι σημαντικό, σαν θέμα αυτό κάθε αυτό, αλλά σαν ε, μέσο επίσης. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε με τις τρίτες χώρες. Μιλούσα με βουλευτές από το Κοινοβούλιο του Μαρόκου και με τα χαράς μπορέσα να τους πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τονίζει τη σημασία που έχει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντί να παίζει το ρόλο δασκάλου εναντί τρίτων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδεικνύει ότι είμαστε πρόθυμοι να ελέγχονται οι πράξεις μας και να ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα εξωτερικό. Και τώρα έχουμε και επίτροπο, ο οποίος είναι υπεύθυνο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο τομέα. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα του όγκου, του φόρτου εργασία που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο εργασία και υποθέσει που πρέπει να διεκπαιρεωθούν και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχουν και πρωτόκολλα σχετικά με βασανιστήρια, ρατσισμό και άλλα θέματα και δικαστική απόδοση που θα πρέπει να προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η υπογραφή της Συμφωνίας Ένταξης Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών είναι κάτι περιορισμένη σημασία, γιατί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάντα ήταν το πρότυπο στην Ευρώπη και ε, περιλαμβανόταν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στις πολιτικές των διαφόρων κρατών μελών. Επίσης, είναι γεγονό ότι θα μπορούσε να υπήρχε και κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την ομολογία που θα διαμορφωθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότατα τόσο ώστε να αποφευθούν σφάλματα. Το, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό το δικαστήριο θα αποκτήσει πυγμή έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Επίσης αξίζει να σκεφτούμε το πώς τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά δικαστήρια λειτουργούν. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Λοιπόν, για 1,5 λεπτό από τους μη η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι δεν κατανοώ ως ε, άτομο που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ποια είναι η προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την προστασία των βασικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο του Στρασβούργου όταν ήδη υπάρχουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, δεν είναι οι δήμονες, μπορεί να παρεξηγήσουν ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν νομικά εργαλεία. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελεί ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα της, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όταν υπάρξει μια προσβολή λοιπόν των δικαιωμάτων ενός πολίτη μπορεί αυτός να στραφεί στο δικαστήριο του Στρασβούργου το οποίο θα του δώσει νομική θεραπεία. Αυτή είναι λοιπόν μια δυνατότητα και γνωρίζουμε όλοι η οποία υφίσταται ήδη σήμερα. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αυτή τη στιγμή αυτήν την δυνατότητα. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή να προσφύγει στο ΕΔΑΔ αν δεν τον ικανοποιήσει η δικαιοσύνη της χώρας του. Ποια είναι η προσθέμενη αξία λοιπόν Ευχαριστώ πολύ, <clears throat> κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι έχουμε σημαντικές στιγμές τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα στη συζήτηση. Υπήρξαν εμπόδια τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν για την προσχώρησή μας στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για νομικούς λόγους και τώρα συζητούμε για το, την εντολή διαπραγμάτευση της Κομισιόν ώστε μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλος της σύμβασης αυτής. Το έγγραφο της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δίνει τη δυνατότητα προστασία του πολίτη έναντι του κράτους μέλους του και είπε σωστά η κυρία Επίτροπος ότι από το Δεκέμβριο η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι νομικά δεσμευτικό και είναι το έγγραφο αναφοράς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη της Λισαβόνα. Η, σύμβαση, η παρουσία της σύμβασης αυτής ενισχύει την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Χάρτα ενισχύει τη Σύμβαση ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το πιο σημαντικό λοιπόν ερώτημα είναι ποια είναι η προσθέμενη αξία για τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έποψη αυτή θέλω να δώσω στη γνωμοδότησή μου μια απάντηση η οποία ενεκρίθη από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να πράξουν στις διαπραγματεύσεις όλα τα απαραίτητα ώστε να γίνει πραγματικά με τρόπο η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προκύψει μια προσθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη χωρίς να δημιουργήσουμε ιδιαίτερα <clears throat> φιλόδοξες και υπερβολικά φιλόδοξες μάλλον προσδοκίες. Υπάρχει το ερώτημα της σχέσης των δικαιοδοσιών των δικαστηρίων του ΕΔΑ δηλαδή και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι <clears throat> η μεταρρύθμιση του ΕΔΑΔ μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της ε, προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο, για ένα πρωτοφανές αν θέλετε εγχείρημα και πείραμα αλλά αυτό δεν θα πρέπει να θέσει ένα αμφιβόλο αυτά τα οποία ήδη λειτουργούν θετικά στο ΕΔΑΔ. Επίσης αυτή η προσχώρηση θα είναι επιτυχής αν μπορούν τα άτομα να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν κατά των θεσμικών οργάνων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικαιοδοσία. Δεν πρέπει λοιπόν να πετάξουμε το βρέφο μαζί με τα ύδατα του μπάνιου, του ιδίου αυτού βρέφους. Ζούμε μια ιστορική στιγμή, νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει το σωστό δρόμο και θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν και το Συμβούλιο να τηρήσουν και να υποστηρίξουν τις ε, προσδοκίες όλων και να ακολουθήσουν αυτή την εντολή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπένοβα. Θέλω να σας πω όμως... Θα ήθελα... Ότι είσαστε, είσαστε η πρώτη συνάδελφος από την Ουγγαρία που λαμβάνει το λόγο και θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Πάλσμιτ έχει γίνει πλέον βουλευτής του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Μας λείπει τα μάλα, θα ήθελα να του, διαβε... να διαβάσετε τα συγχαρητήριά μας και είμαστε σίγουροι ότι θα παίξει πλήρως το ρόλο του ως πρόεδρος του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Φλασικόβα Μπένοβα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους Ούγγρους συναδέλφους. Και τώρα πίσω στο θέμα μας. Παρόλο που όλα τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη στην σύμβαση. Η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι απλώ μια νέα διάσταση που προστίθεται όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το τονίζω αυτό, θα είναι νομικό και πολιτικό μήνυμα το οποίο θα ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ευρώπης. Μαζί με την προσχώρηση, τη συμφωνία προσχώρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει την κοινωνική χάρτα. Αυτό θα ήταν ένα γεγονός ευπρόσδεκτο, ένα σωστό βήμα. Η πολιτική προσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης δημιούργησε κάποια ερωτηματικά, καθώς και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά και η διαδικασία, Επίτροπε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας, μεν, και ευχαριστώ και το Συμβούλιο για τα όσα έκανε. Θεωρώ όμως, δε, ότι αυτή η διαδικασία θα είναι δύσκολη και πολλή δουλειά θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μιγάλσκι. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μία από τις πιο ευγενείς πτυχές ε, του όλου θεσμού, αλλά μου φαίνεται ότι μιλάμε υπερβολικά πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των δικών μας πολιτών. Η κυρία Μπένοβα το είπε, η κυρία Βίκστρομ το είπε. Νομίζω ότι δεν κάνουμε αρκετά από αυτά που ανέφερε η κυρία Χάουταλα, δηλαδή να διασφαλίζουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων εκτός των ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αρκετά στον τομέα αυτό. Επικροτώ την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση. Πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνέπεια όσον αφορά την ε, εφαρμογή της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν θα πρέπει να περικόπτονται οι ελευθερίες όταν θεσπίζονται νέα δικαιώματα. Είναι θέμα σημαντικό, όχι μόνο φιλοσοφικό και οι βουλευτές και οι δικαστές θα πρέπει να το γνωρίζουν καλά. Ένα λεπτό για την κυρία Βέρθμαν. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρο 6, προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που σημαίνει ενίσχυση ε, του συστήματο ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η προσχώρηση σε αυτό το νομικό σύστημα θα ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έχουν κερδίσει ένα επιπλέον νομικό μέσο σε περίπτωση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι πολύ θετική, ε, διότι έτσι ε, ενισχύεται η συνείδηση, των, η συνείδησή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυξάνεται η προστασία. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ο κύριος Τσαρκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές μας και την Κίνκα Γκάλ και τον Ραμόν Χαουρεγγί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο σκληρό αλλά απαραίτητο έργο σας. Όταν μιλάμε για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούμε εδώ και 10 χρόνια. <clears throat> Πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει ανταγωνισμό μεταξύ των δύο δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Θα υπάρξουν, λένε πολλοί, πολλά προβλήματα σε σχέση με τι δικαιοδοσίε αυτών των δικαστηρίων. Η αυτονομία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο. Αλλά αυτό το οποίο αναμφιβόλα θα επιτευχθεί είναι ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα δύο αυτά δικαστήρια μπορούν να παίξουν ένα συμπληρωματικό ρόλο. Θα πρέπει να πράξουμε όλα τα απαραίτητα για να έχουμε μια καθαρά ιεραρχική σκέψη αντί να δεχτούμε την διασταύρωση των νομολογιών των δύο δικαστηρίων. Όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ακολουθεί την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και Τούμπαλιν, έτσι τα δύο συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός και δεν θα υπάρξει ασάφεια του δικαίου. Στην πρόσφατη απόφαση Βόσφορους η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος το ΕΒΔΑΔ μάλλον είπε ότι δεν υπάρχει λόγο να επανεξεταστεί το θέμα αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ήδη ένα επαρκέ επίπεδο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ερώτημα λοιπόν εγείρεται γιατί χρειαζόμαστε αυτή την προσχώρηση και τέθηκε από του συναδέλφου μα εδώ. Το χρειαζόμαστε όχι μόνο λόγω συμβολικού νοήματο κάτι το οποίο είναι αφεαυτού σημαντικού, αλλά γιατί με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε το σύστημα προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, θα αυξήσει την αξιοπιστία του ενώπιον των πολιτών και θα καλύψει τους πολίτες όχι μόνο εναντί των κρατών μελών αλλά και εναντί της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Όταν δεν υπάρχει αποτελεσματική νομική θεραπεία, όταν παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να προσφύγει ο πολίτης εναντίον ενός σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα θα καλύπτεται αυτή η ανάγκη. Θα μας δώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή η προσχώρηση και για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το σύστημα θα πρέπει να έχουμε και ένα πνεύμα πιστό στο πνεύμα. Γι' αυτό ε, πρέπει να αποφασίσουμε να μην φέρνουμε στο δικαστήριο του Στασβού προσφυγές κατά μεταξύ κρατών μελών και να δεχόμαστε τις αποφάσεις του και να τις εφαρμόζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχει δημιουργήσει μια Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως φοιτητή εγώ διάβαζα τα άρθρα του Βάιλερ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είπε ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε σε σχέση με τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά αν δεν υπάρξει μια παρακολούθηση και εφαρμογή από την Κομισιόν, δεν θα επιτύχουμε ποτέ. Χάρη σε εσά λοιπόν έχουμε αυτή την πορεία που ελπίζουμε ότι θα καρποφορήσει και θα δώσει καλύτερη προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ό,τι τώρα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο λεπτά στον κύριο Σιόγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόσθεση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και έτσι ε, κάνει ένα ε, περαιτέρω βήμα στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ε, και έτσι επιβεβαιώνει και την αξιοπιστία της απέναντι στις τρίτες χώρες όπου προσπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την πράσινη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα ε, να καλέσω την ε, Κομισιόν να κάνει και τα περαιτέρω βήματα και να πάρει μέτρα για βελτίωση της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι θα γίνει χώρος ε, ελευθερίας, ε, ασφάλειας και δικαιοσύνης με τα επιτεύγματα αυτά στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει να αναφέρουμε τον ε, χάρτη των εθνοτικών ε, και περιφερειακών μειονοτήτων. Θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα το, την Συμφωνία Πλαίσιο για την προστασία των εθνοτικών μειονοτήτων. Η συμφωνία αυτή ε, θεσπίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ε, μειονοτήτων. Όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης και τα περισσότερα από αυτά έχουν υπογράψει και επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση με την ε, υιοθέτηση των συμφωνιών αυτών που χρησιμοποιούνται ευρέω, μπορούμε να ενισχύσουμε ε, το σύστημα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τελευταίο λοιπόν ομιλητή κλείνουμε τον κατάλογο αυτών που ήταν εγγεγραμμένοι ε, ατομικά για να λάβουν το λόγο και περνάμε τώρα στο, στην θύρα οφθαλμών στη διαδικασία Catch the Eye όπου έχουμε έξι άτομα που ζήτησαν τον λόγο ο κανονισμό λέει μπορώ να δώσω το λόγο σε πέντε, α είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι. Παρακαλώ όμω να παραμείνετε στα πλαίσια ενό λεπτού, γιατί αλλιώ θα πρέπει να σα κόψω το λόγο. Η κυρία Μπασέσκου είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε. Με την θέση εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας έχουμε στα χέρια μας μια εγγύηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το Δικαστήριο του Σασβούρου θα εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών έναντι των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τα κράτη-μέλη έχουν ε, εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικούς τομείς αρμοδιότητας. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε περιστολή των δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαστήριο του Λουξεμβούργου εξακολουθεί να είναι το ανώτατο δικαστήριο για όλε τι ε, ε, αγωγέ και προσφυγέ που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του κοινωνικού δικαίου. Εμείς έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει την ε, απόφαση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 1993 και υπάρχει στο Σύνταγμα της Ρουμανίας ένα άρθρο που λέει ότι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διεθνείς δικαίω. ε, συμφωνίες έχουν προτεραιότητα εναντίον του εθνικού δικαίου. Ο, ο κ. Σταμπατζή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο λειτουργεί πολύ καλά και το οποίο έχει ένα σωστό επίπεδο ελέγχου ε, είναι τώρα τμήμα και της ε, ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εδρεώσει το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πολύ καλά, αλλά δεν έχει το πολιτικό βάρος και ανάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Θα ήθελα να τονίσω αυτό γιατί και η κυρία Γκάλα αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Αναφέρθηκε στο θέμα της ε, υπεροχής της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εδώ πρόκειται <clears throat> μάλλον τη υπεροχή του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Εδώ πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ε, μειονότητες. 6 με 8% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες εξάλλου. Ευχαριστώ, λέει ο Έχετε το λόγο, θέλω συγχαρώ τον κύριο Χάουρεγγι για το τόσο σημαντικό έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρα η κυρία Μπιλμπάου και που καλύπτει τις θεσμικές πτυχές της προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ και πολλές δεκαετίες το Κοινοβούλιο και η Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σύμβαση. Τώρα με 27 μέλη κανεί δεν διαμφισβητεί την ανάγκη αυτή τη προσχώρηση. Αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει και βάση ταυτότητα και πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε κρίσει να αντιμετωπίσουμε και πολιτικά προβλήματα και όχι μοναχά οικονομικά. Το να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίε σε όλε τι συνθήκε χωρί κανένα δισταγμό, αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε και τη δημοκρατία, την πρόεδρο και σημαίνει ότι θέτουμε στο περιθώριο οποιαδήποτε έκφραση βίας ή εφαρμογή αυταρχικών τάσεων. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ακριβώς και ο στόχος, της, το αρχικό νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή πρέπει να είναι η πορεία μας και ζητώ από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν αυτή την ε, κίνηση και θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα στην Ελλάδα. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ποιος? Κάποιος Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών είναι μια είναι ένας από τους πυλώνες ε, του ε, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ε, έχει εμπνεύσει τις αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση κατά την ίδρυσή τη. Επί πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε τη δουλειά του ε, ε, υπερασπιζόμενο τους αδύναμους και τους διοκόμενους. Ωστόσο, μια σειρά αποφάσεων έχουν οδηγήσει σε αμφιβολίες. Πέρσι, ακούστηκε ένα κύμα αντίθεσης σε μια απόφαση ε, που απαγόρευε τους ε, σταυρούς δημοσίως. Πιστεύω ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην σύμβαση αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στο ξεκίνημα μιας συζήτησης για να διασφαλίσουμε Ε, την αποφυγή αυτή της ε, λάθο ερμηνείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέλλον. Ο κύριος Καλινόφσκι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει υιοθετήσει προτάσεις ψηφισμάτων που καταδικάζουν τις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ίδια τα κράτη-μέλη μας. Πρόσφατα, η Επιτροπή Ηθικής της Λιθουανίας καταδίκασε τον συνάδελφο Τομασέφσκι επειδή έθεσε ερώτημα ε, ε, προς τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω αν η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση θα βοηθήσει, διότι χρειαζόμαστε πολύ υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων από ό,τι έχουμε στην σχετική λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Θέλω και εγώ καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για την απώλεια τριών Ελλήνων πολιτών σήμερα για τον χαμό τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο ειρηνικών διαδηλώσεων ε, των Ελλήνων πολιτών για ένα καλύτερο μέλλον. Κάποιοι λειτουργώντας περιθωριακά, κάποιοι λειτουργώντας αντιδημοκρατικά, αφαίρεσαν τόσο άδικα τις ζωές των συμπολιτών μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πραγματικά τραγική ηρωνία να συζητάμε σήμερα για την ε, ενίσχυση και την ευάνθηση στο πλέγμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών με την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρίε και κύριοι, όσο και να δουλέψει αποτελεσματικά το Δικαστήριο του Στρασβούργου, πρέπει να ξέρουμε ότι για να ενισχύσουμε την ιδέα της Ευρώπης, μια Ευρώπη των αξιών, μια Ευρώπη με κέντρο τον άνθρωπο, αυτό που πρέπει να είναι η κορυφαία αναφορά όλων μας είναι η αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλληλεγγύη ε, μεταξύ των λαών, αλληλεγγύη τόσο έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και με την παρέμβαση των συναδέλφων που έλαβαν το λόγο σε ό,τι αφορά την οφθαλμοθυρική διαδικασία Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να δώσουμε στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και μετά στην εκπρόσωπο της Κομισιόν για να κλείσει η συζήτηση σε αυτό το σημείο. Κύριε Λόπες Καρίδο, έχετε το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι σχεδόν οι βουλευτές οι οποίοι έλαβαν το λόγο υπεστήριξαν την ε, υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμφωνούμε μαζί τους και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στις δύο παρεμβάσεις οι οποίες έδειχναν κάποιες αμφιβολίες ή ακόμα και κάποιες αντιρρήσεις στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θεωρώντας ότι ήταν αυτό κάτι το επικίνδυνο, όπως είπε ο κ. Ζιόμπρο, για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι ήταν κάτι το περιττό, όπως είπε η οτι ηταν κατι το πέριτο, οπως ειπε η κ. μορβαη Θέλω να απαντήσω και στους δύο βουλευτές. Το επιχείρημα του κ. Σιόπρο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Διότι το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν μπορεί να υπησέλθει σε αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και ο στόχος του. Το πρωτοκόλλο 8 της Συνδίκης της Λισαβόνας επίσης καθιστά σαφές ότι με τον τρόπο αυτό δεν τροποποιούνται καθόλου οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ακόμα και τα θέματα τα οποία εξετάζονται από την ομάδα εργασίας <clears throat> για το μηχανισμό της συνεναγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν υπάρχει μια προσφυγή κατά ενός κράτους μέλους στο δικαστήριο του Στρασβούργου εναντίον ενός κράτους μέλους να θεωρείται συνεναγόμενη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό έχει ακριβώς σαν στόχο να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα αφού εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα προηγουμένως. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο επεξεργάζεται η ομάδα αυτή εργασίας για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι υπήρξε προηγουμένως εξάντληση ε, ενδίκων μέσων. Το ΕΔΑΔ λοιπόν απλώς μπορεί να ε, να εξασφαλίσει, να διαπιστώσει την, πα, την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όχι, αλλά δεν μπορεί να έχει την τελική δικαιοδοσία. Για την κυρία Μορβάη τώρα. Ε, λέει ότι εγώ μπορώ να προσφύγω στο ΕΔΑΔ εναντίον μια απόφαση στο κράτο μέλο μου. Γιατί πρέπει να προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι σαφέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σειρά αρμοδιοτήτων που ξεπερνούν τι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες και επίσης έχει αρμοδιότητες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο θεσμός ο οποίος παίρνει αποφάσεις μέσω κανονισμών, μέσω οδηγιών, μέσω αποφασίσεων, μέσω αποφάσεων νομικού χαρακτήρα που μπορούν να θίξουν τα δικαιώματα των πολιτών, μπορούν να θίξουν τη Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτό η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μεγαλύτερες εξουσίες καθιστά απαραίτητο και γι' αυτό το δεσπίζει και η Συνδίκη της Λισαβόνας ότι όπως και τα κάτι μέλη που προσχώρησαν στο, στη Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΔΑΔ, τότε επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να υπόκειται στην, ομο, στην δικαιοδοσία, στην δοσυνδικία καλύτερα, του ΕΔΑΔ. Και η η λειτουργία του ΕΔΑΔ ήταν πάντα πάρα πολύ σημαντική για την προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η Σύμβαση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που είναι το κείμενο το οποίο εφαρμόζει το ΕΔΑΔ είναι ένα κείμενο του 1950 πριν από τη Συνδίκη της Ρώμης. Είναι και αυτό μια σύμβαση που έγινε στη Ρώμη και συμπληρώθηκε με μια σειρά πρωτοκόλλου. Παρ' όλα αυτά έχει δημιουργηθεί μια πλούσια νομολογία η οποία έχει επηρεάσει την ομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων και των συνταγματικών δικαστηρίων των κρατών της, Ευρω... της Ευρώπης και έχει δημιουργήσει ένα, μια κοινή περιουσία νομική που παίζει σημαντικό ρόλο για την ερμηνεία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταξύ του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου. Για όλου αυτού του λόγου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση αυτό θα προστατεύσει όχι μόνο κατά τους πολίτες από τα κράτη-μέλη, αλλά και τους πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι πολίτες, δεν είναι ηθαγενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η σύμβαση αυτή προστατεύει όλα τα άτομα τα οποία βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών και επομένως το μέλλον αυτό θα καλύπτει και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν και πολίτες που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής λοιπόν εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Θέλω επομένω να τονίσω ότι μας ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει μια συνένεση για την ανάγκη να προχωρήσουμε με την ε, ε, εκπλήρωση αυτής της εντολής <clears throat> που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όπως είπε και ο κύριος Χαουρεγγί θα λάβει χώρα μια συζήτηση στην Ορομέλεια το Μάιο για το θέμα αυτό και θέλω να το συγχαρώ και αυτόν και τους υπόλοιπους εισηγητές για τα θέματα αυτά στη Συνταγματική Επιτροπή, Πρέντα και Γκάλ και πιστεύω από την πλευρά της Ισπανικής Προεδρίας θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η έγκριση αυτής της εντολής επί τη βάση του κειμένου της Κομισιόν που φυσικά η Κομισιόν θα πρέπει να είναι ο διαπραγματευτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών των θεμάτων εσωτερικών και δικαστικών θεμάτων της 4ης Ιουνίου προσεχώς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκαρίδο και θα κλείσουμε με την παρέμβαση της Επιτρόπου της Αντιπροέδρου κυρίας Ρέντινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω λέγοντας πόσο συμφωνώ με τα όσα εξέφρασε μόλις τώρα εν ίδια απαντήσεως η Ισπανική Προεδρία εν ίδια απαντήσω ερωτήσεις των βουλευτών. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν, δεν θα έλεγα ακριβώς τα ίδια. Επιτρέψτε μου απλώς να ευχαριστήσω τους βουλευτές που πήραν το λόγο με επικοδομητικό τρόπο για να υπογραμμίσουν τη σημασία που έχει το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελούν τη βάση της Ένωσής μας και η ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για κάθε πολίτη μπορεί να αποτελεί μόνο πρόοδο σχετικά με αυτό που θεωρούμε πραγματικές αξίες της Ευρώπης μας. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος τους δύο συγητές που έκαναν πολύ σημαντική δουλειά. Έτσι το Κοινοβούλιο συμφώνησε επί της βασικής εντολής. Η βασική εντολή, όπως αναφέρθηκε, είναι απλώς η αρχή, διότι πρέπει να διαπραγματευτούμε. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο και όταν περατωθούν οι διαπραγματεύσεις τότε έχουμε τη διαδικασία επικυρώσεως που πρέπει να ξεκινήσει. Λοιπόν, Πρόεδρε, προβλέπω ότι πολύ συχνά θα πρέπει να επανέλθω με χαρά μου στο Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να ενημερώσω σχετικά για το πού βρισκόμαστε, πώς προχωράμε, πού βρίσκονται τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις και πιστεύω ότι οι βουλευτές θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να πετύχουμε τον κοινό στόχο που είναι μια Ευρώπη αξιών και δικαιωμάτων. Θα είναι ευχαρίστηση για μας, αλλά μάλλον θα είναι και κοινή ευχαριστήση μαζί με την κυρία Αντιπρόεδρο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, της δηλώσης του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε σχέση με τα